με το νομοθέτημα για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές εταιρείες θα μπορέσει και ο ίδιος να τοποθετηθεί προσωπικά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τελείωσε αυτή η συζήτηση. Τώρα με βάση την ημερήσια διάταξη περνάμε στην προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τον καονισμό σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της καταγωγής ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Το λόγο έχει καταρχήν ο κύριος Μορέιρα, που είναι ένας από τους συντάκτες, και μετά ο άλλος συντάκτης. Ενάμιση λεπτό. μισή λεπτά, συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι από τους ε, συνυπογράφοντε τη προφορική ερώτηση ε, και να πω και σε μένα να την παρουσιάσω στην Ολομέλεια. Στα τέλη του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ένα σχέδιο κανονισμού για την εισαγωγή υποχρεωτικού συστήματος ε, ε, προέλευσης για κάποια εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες. Στόχοι της πρώτης αυτής ήταν πρώτον αποφυγή ψευδών ή παραπλανητικών δείξεων προέλευσης, ενημέρωση καλύτερη του καταναλωτή για την καταγωγή κάποιων προϊόντων, ε, ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών προϊόντων έναν των προϊόντων τρίτων χωρών όπως Καναδάς Κίνας, Ιαπωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών που ήδη επιβάλλουν ε, ένδειξη προέλευσης στα εισαγόμενα προϊόντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα ανέκαθεν υπέρ ενό υποχρεωτικού καθεστώτος ε, επισήμανσης της ε, προέλευσης, όπως αναφέρουν τα ψηφίσματα του 2006 και του 2009. Τον Οκτώβριο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις νέες του νομοθετικέ αρμοδιότητες σε εμπορικά ζητήματα που απορρέουν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, εγκρίναμε μία θέση σε πρώτη ανάγνωση για το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την αναφορά χώρας προέλευσης για ορισμένες αγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα. Μάλιστα το αποτέλεσμα ήταν 529 ψήφοι υπέρ, 49 κατά και 44 αποχές. Στη συνέχεια και παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο δεν κατάφερε να καταλήξει εκείνη η θέση, μπλοκάροντα ουσιαστικά την νομοθετική διαδικασία. Πρόσφατα, σε μια απρόσμενη τροπή των γεγονότων, η Επιτροπή ανήγγειλε θα αποσύρει τον ε, κανονισμό κατά τη διάρκεια του 2013 ισχυριζόμενη ότι η απόφαση τη ειδική ομάδα Παγκόσμιου Οργάνωση Εμπορίου σχετικά με την υπόθεση ε, για τα βοηδή και χοιρινά και την ένδειξη προέλευσης άλλαξε ουσιαστικά την ομολογία του ΠΟΕ πράγμα το οποίο καθιστούσε την αρχική πρόταση του κανονισμού Made in μη συμβατή με τις αρχές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Ερωτώ λοιπόν, για ποιο λόγο επιλέγει η Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση αντί να προτείνει τις αναγκαίες αλλαγές ώστε να καταστήσει τον κανονισμό συμβατό με τις αρχές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου συμπεριλαμβανομένης μιας νέας εν ανάγκη νομικής βάσης εάν αυτό είναι ε, που θα εγκριθεί από του συνομοθέτες με την τρέχουσα διαδικασία κατά τη διάρκεια τη δεύτερη ανάγνωση και ενδεχομένω με δια, διαδοχικούς τριμερείς διαλόγους. Δεύτερον, δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι στο πλαίσιο του πνεύματος καλής οργανικής συνεργασία και σεβασμού προ Ευρωπαίου πολίτε, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τη μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θεωρεί λοιπόν ότι θα έπρεπε να είχε διαβουλεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δοθεί επαρκή χρόνο για συζήτηση πριν αναγγείλει την απόσυρση τη πρόταση. Πιστεύει η Επιτροπή ότι η απόσυρση του κανονισμού είναι προ το γενικό συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, ποια στοιχεία τη αρχική πρόταση ή του κειμένου τη πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δεν είναι πλέον συμβατά με τι αρχέ του ΠΟΕ για ποιο λόγο. Σε συνέχεια των αποφάσεων τη ειδική ομάδα του ΠΟΕ και του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ, Ποια είναι η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποχρεωτική ένδειξη τη προέλευση που απαιτείται από πολλέ χώρες, άλλε χώρε εισαγόμενα προϊόντα, όπω η Βραζιλία, ο Καναδά και οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Τέταρτον, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει την ένδειξη τη προέλευση και ω εκ τούτου την χνηλασιμότητα των προϊόντων που εισάγονται από τρίτε χώρε στην ενιαία αγορά, τουλάχιστον για αυτού του τομεί που καλύπτονται ήδη από τον κανονισμό. Και ποιο είναι το προβλεπόμενο σχετικό χρονοδιάγραμμα. τέλο, προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει μια νέα πρόταση για τον ελόγο κανονισμό σύμφωνα με του νέου κανόνε του ΠΟΕ. Και αν ναι, πότε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μουσκαρδίνη για δυόμιση λεπτά. Κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, ακούσατε τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Μορέιρα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι Πρέπει να έχουμε κοινού κανόνες που να του εμεριζόμαστε όλοι. Η ελευθερία ε, του εμπορίου και του ανταγωνισμού θα πρέπει να εξασφαλιστούν, ιδίω στο εσωτερικό του ΠΟΗ. Δεν μπορεί να υπάρχουν καταναλωτές και παραγωγοί τάξης Α και τάξης Β ανάλογα με τη χώρα ή ανάλογα με την Ήπειρο στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται. Έχουμε σημαντικούς ε, εταίρους, εμπορικούς εταίρους, Κίνα, ε, Βραζιλία, ΗΠΑ, που επιβάλλουν ε, την υποχρεωτική ένδειξη καταγωγής σε ορισμένα προϊόντα που έρχονται από το εξωτερικό, τότε και εμείς ως Ευρώπη έχουμε το δικαίωμα να έχουμε αντίστοιχους κανόνες. Και επομένως και το καθήκον να έχουμε ένα κανονισμό για την ε, σήμανση κάποιων προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό όπως ψήφισε το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο ε, του 2010 σε πρώτη ανάγνωση. Ή θα έχουμε αυτόν τον κανονισμό ή τότε θα πρέπει να ζητήσουμε από τον ΠΟΕ να παρέμβει, ούτως ώστε να καταργήσει τους κανόνες της χώρες που υπάρχουν αυτές. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορούμε να έχουμε μια παγκόσμια αγορά σωστή, εάν κάποιοι ευνοούνται και κάποιοι άλλοι όχι. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι σωστή απέναντι στους δικούς της καταναλωτές, πολίτες και παραγωγούς αν δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα μαζί με τα καθήκοντα. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν με τα λόγου γνώσεως. Και το ευρωπαϊκό σύστημα, ε, το ευρωπαϊκό βιομηχανικό σύστημα που είναι η σπονδυλική στήλη της, του ανταγωνισμού μας θα πρέπει να λειτουργεί με βάση κάποιους ε, προβλέψιμους κανόνες. θα πρέπει να έχουμε και εμείς τα ίδια δικαιώματα με αυτά που έχουν οι καταναλωτές και οι εταιρείες στην Κίνα, Βραζιλία, ΙΠΑ κτλ. Θα πρέπει η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συζητήσουν πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Εμείς δεν έχουμε την αλαζονία να πιστεύουμε ότι αυτό που ψηφίσαμε είναι θέσφατο και ότι δεν αλλάζει. Απλώς ζητάμε να μην υπάρχει αλαζονία ούτε από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από πλευρά Συμβουλίου. Αλλά αυτό συνέβη σε αυτή την αξιολύπητη κατάσταση όπου η Κομισιόν δεν θεώρησε καν ότι είναι σωστό να μας ενημερώσει εγκαίρως. Να ενημερώσει δηλαδή την καθήλυνα αρμόδια ε, κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι η Επιτροπή Εμπορίου. Θα έπρεπε με μέσω μια άτυπη συνάντηση μεταξύ των τριών ε, θεσμικών οργάνων να δούμε ποιοι συμβιβασμοί θα πρέπει να προωθηθούν για να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση για να ξεκαθαριστούν τα θέματα γιατί το πρόβλημα είναι ακαθόδε. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Δεχούχτ έχει το λόγο. Thank you, uh, Madam Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εταιρείε ε, μπορούν να ορίσουν την προέλευση των προϊόντων. Εκείνοι που κάνουν την πρόταση λεγόμενη made in ε, φιλοδοξούν στη σήμερα των προϊόντων των βιομηχανικών. Ξέρουμε ότι ε, το Κοινοβούλιο προς τη μεγάλη σημασία στην προέλευση και τη σήμανση της προέλευσης και μάλιστα φάνηκε αυτό και από την υποστήριξη της αντίστοιχης έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ε, προωθηθεί αυτή η νομοθετική πρόταση και λαμβάνει υπόψη τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Επτά έτη, επτά έτη μετά την κατάθεση της ε, πρότασης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Δεν έχει προχωρήσει υπόθεση από την ε, ψήφισε στο Κοινοβούλιο και μετά ότι υπάρχει τέτοια προοπτική μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Επιπλέον, ε, σύμφωνα με πρόσφατε αποφάσει του ΠΟΕ, υπάρχουν μεγάλε ανησυχίε για το κατά πόσο η πρόταση αυτή συνάδει με ε, του κανόνε του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Για πρώτη φορά ορίζεται ότι υπάρχει τέτοια συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια του εμπορίου. Στον ΠΟΕ. Και είναι αυξημένο ο κίνδυνος για την πρόταση Made in να επιβάλλεται μόνο σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και όχι στα ε, κοινοτικά προϊόντα. Επίσης, από τότε που ξέσπασε η κρίση, εστιάζεται η πρόταση στις εισαγωγές και είναι πιο επίμαχη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους ισχυρότερους συνήγορους ε, ε, κατά του προστατευτισμού. Θα πρέπει λοιπόν πολύ προσεκτικά να τα εξετάσουμε και το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πρόγραμμά της για το έτος 2013 έχει συμπεριλάβει ε, την απόσυρση ε, της πρότασης. Είναι πρόθεσή μας. Είμαστε μεσούσει τη ε, θεσμική διαδικασία, Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν και ενδεχομένω να αποφασίσει την απόσυρση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητήθηκε στην Επιτροπή ε, διεθνούς εμπορίου και μάλιστα στις 10 Ιανουαρίου έγινε και μια αντίστοιχη τεχνική σύσκεψη. Σε ό,τι αφορά τη σήμανση προϊόντων ε, και των αντιστοίχων αγορών υπάρχει αυτό σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά ε, όλα αυτά τα συστήματα διαφέρουν μεταξύ τους και είναι προγενέστερα της πρόσφατης απόφασης του ΠΟΕ. Ε, δεν έχουμε λάβει όμως ε, καμία αναφορά για μεγάλα εμπόδια που γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς λόγω αυτών των ε, συστημάτων. Αν κάτι τέτοιο υποπέσει την αντίληψή μας θα το εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Έχουμε λοιπόν και διεθνείς υποχρεώσεις όπως ορίζονται στις πρόσφατες αποφάσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι δεν μπορεί να προωθήσει αντίστοιχη νομοθεσία για την προέλευση εισαγωμένων ειδών ε, διαφορετική από αυτή που υπάρχει στην πρόταση η οποία αυτόν τον καιρό ε, έχει οδηγηθεί σε αποτελμάτωση. Η αρχική πρόταση επιβάλλει τη σημασία ε, προέλευσης όχι μόνο για εισαγόμενα προϊόντα αλλά και με μια ετικέτα Made in European Union. Αυτό αλλάζει όμως το πεδίο εφαρμογή της πρότασης άρα χρειάζεται νέα πρόταση σε διαφορετική νομική βάση. Δεν πιστεύω κύριε Μορέιρα ότι αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παρούση διαδικασίας. Αυτό σημαίνει και χρειάζεται μελέτη αντικτύπου για να δούμε αν μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα ικανοποιεί ε, τους όρους της συνθήκης. Υπάρχει ε, και αίτημα του κλάδου και ε, προσδοκία των καταναλωτών προς την κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε τώρα επιπλέον κόστος στις εταιρείε μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολουθεί αυτή την οδό. Είτε θα Συνεχίζει να το εξετάζει ο αρμόδιος επίτροπος ε, Ταγιάννη, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, θα το ε, εξετάσει. Ας επανέλθουμε όμως ε, στα ουσιαστικά και το υπόβαθρο. Τι μας ενδιαφέρει, να υπάρχει ένα πλαίσιο ίσων όρων παιχνιδιού για τις εταιρείες μας, προστασία από ψευδή και πλαστή ένδειξη προέλευσης και ενημέρωση των καταναλωτών. Πρόσφατες μελέτες ε, για ε, τη γλωστοεφαντουργία και τα δερμάτινα δείχνουν ότι στην αγορά αυτό δεν είναι ε, πρώτος προτεραιότητα και σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή θέλει να ενισχύσει την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές ε, πρακτικές με μέτρα που περιλαμβάνουν νομοθετική πρόταση για την εποπτεία και παρακολούθηση της αγοράς τέτοιων προϊόντων για βελτίωση του ελέγχου και επιβολή του στην Ένωση. Η νομοθετική πρόταση για την γενική ασφάλεια προϊόντων και πολιετές πρόγραμμα για ε, επιτήρηση της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται αλλά έχει προβλήματα και ε, ε, πόρων και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προαχθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη. Απαντώ στις ερωτήσεις των συντακτών λέγοντας ότι Έχουμε ξεκαθαρίσει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι προτιθέμεθα να αποσύρουμε την ελόγω πρόταση. Έχει ενημερωθεί μέσω του Προέδρου της Επιτροπή Εξωτερικού Διεθνούς Εμπορίου και έχουμε και το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2013 και θα ενημερώσουμε και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, για τις προθέσεις μας και τα σχέδιά μας. Αυτό εντάσσεται πλήρως στη συμφωνία πλαίσιο. Ε, το Κοινοβούλιο έχει την ευκαιρία να κάνει τις ε, παρατηρήσεις του και να εκφράσει την άποψή του πριν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε να αποσύρει αργότερα την άνοιξη την πρόταση είτε να ακολουθήσει διαφορετική τακτική. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ το λόγο έχει ο κύριος Κασπάρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά την άποψή μου, περί τίνος πρόκειται σήμερα. Δύο ζητήματα. Είναι το θεσμικό αφενός, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ και μήνες, για να μην πω χρόνια, μας έχει κάνει ε, νομοθετική πρόταση. Σε πρώτη ανάγνωση το ψηφίσαμε και με μεγάλη πλειοψηφία και το Συμβούλιο, το οποίο απουσιάζει και σήμερα, περιμένει δύο χρόνια και αδρανεί. Και τώρα συμφωνούμε ότι η αδράνεια του Συμβουλίου και αυτή η ολιγορία, η ο σύνομοθέτης δεν έχει αναλάβει καμία πρωτοβουλία, μηδέν. Ε, αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται. Ε, είναι απαράδεκτα. Και το δεύτερο, κύριε Επίτροπε, εσεί ανακοινώσετε στο πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλετε να αποσύρετε την πρόταση. Εγώ θα επιθυμούσα ε, σύμφωνα με τα δεδομένα, δεν, ε, μπορεί να μην μου άρεσαν όλε τι λεπτομέρειε, αλλά η πρώτη ανάγνωση έχει ολοκληρωθεί. Θα προτιμούσα να προσπαθήσετε μαζί μα να κάνετε την πρόταση αυτή συμβατή με τον ΠΟΕ αντί να την αποσύρετε. Ε, πολλά προϊόντα ήδη έχουν σήμανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που εισάγονται εννοώ. Και κατανοώ ε, και τους καταναλωτές. Μπορεί να είναι και λίγοι που να ενδιαφέρονται, αλλά σήμερα ο κόσμος είναι παγκοσμιοποιημένο. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ε, στον καταναλωτή ε, που έχει κατασκευαστεί ε, ένα προϊόν όταν γίνεται σε 30, 40, 50 χώρες. Υπάρχουν προϊόντα πολύ περίπλοκα με προμηθευτές, με υπεργολάβους. Πού θα το γράφει στο Made in. Αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται και ο καταναλωτής. Αν δεν έχουμε καμία ρύθμιση τότε έχουμε πάρα πληροφόρηση. Ε, των καταναλωτών. Θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε γι' αυτό και να δούμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε, ενδεχομένω μια νέα πρόταση που επιθυμώ εγώ. Ευχαριστώ. του σοσιαλιστές, ο κύριος Σούστα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και άλλοι συνάδελφοι υπενθύμησαν το θεσμικό γόρδιο δεσμό που προήλθε από την απόσυρση της πρότασης της Κομισιόν. Εμείς είχαμε χαιρετήσει θετικά, κύριε Επίτροπε, τη δική σας πρωτοβουλία πριν από τρία χρόνια να ξαναπροτείνετε μετά από τη θεσμική αλλαγή που συνέβη με τη συνθήκη της Λισαβόνας τον καονισμό για το Made in και να εμπλέξετε το Κοινοβούλιο με ενεργό τρόπο ε, και να το καταστήσετε συνομοθέτης. Με δυσκολία καταλαβαίνουμε για ποιους λόγους πραγματικά αλλάξατε θέση. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι από τη μία πετάτε έξω το κοινοβούλιο, το οποίο όχι απλώς ένα απλό ψήφισμα, αλλά με νομοθετικό τρόπο εξέφρασε τη γνώμη του. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αυτή η αλλαγή με επίσημο τρόπο ξαναπροτείνατε αυτό που ε, πριν από 7 χρόνια αρχικά είχε ξεκινήσει. Το ψηφίσαμε τον Οκτώβριο του 2010. Αυτή η πρόταση ψηφίστηκε μετά από μια θεσμική συμφωνία μεταξύ Κομισιών και ε, Κοινοβουλίου που επαναδιατύπωσε τις σχέσεις μεταξύ των δύο οργάνων. Το να προσφεύγουμε ε, σε αυτούς που είναι κατά των κάνων αυτών ε, και που ανήκουν στην κοινωνία των πολιτών, αυτό είναι λάθος. Γιατί ούτως ή άλλως τα πιο περίπλοκα συμφέροντα που εκφράζονται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αυτή την ένωση των 500 εκατομμυρίων ε, καταναλωτών, τα εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η βιομηχανία μας που είναι στο κέντρο της κρίσης είναι η μόνη η οποία μπορεί να μας βοηθήσει για να βγούμε από την κρίση και να εξασφαλίσουμε επαρκή επίπεδα απασχόληση ζητούν ακριβώς αυτόν τον κανονισμό. Όχι για προστατευτικούς λόγους, αλλά για να δημιουργηθούν συνθήκες αμοιβαιότητες με τις άλλες χώρες, με τις ξένες χώρες. Χρειάζεται μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Ε, γιατί μην ξεχνάτε τι, ποια πρωτοβουλία έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείε από τη δική του τη μεριά. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αντιπαράθεση μεταξύ Κοινοβουλίου, ε, Κομισιόν και Συμβουλίου. Ε, και να βγούμε από, αυτά τα, από αυτούς τους ύποπτους ε, μηχανισμούς μέσα στους οποίους ε, βουλιάζουμε. Ο κύριος Ρινάλντι για δύο λεφτά. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρουμε ότι με αυτό τον κανονισμό θα δινόταν κάποιες πρωτοβουλίες στους καταναλωτές. Ξέρουμε επίσης ότι αλλού στον κόσμο υπάρχουν τέτοιες διατάξεις. Στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά στο Μεξικό, στην Ιαπωνία κτλ. κτλ. Ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο κατάφερε να πετύχει μια ευρεία πλειοψηφία παρά το γεγονός ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν ουσιαστικές ε, αντιρρήσεις και δισταγμοί από, συναδέλφους ε, που ανήκαν σε, άλλες, σε διάφορες πολιτικές ομάδες ε, και που δεχόταν πιέσεις από κυβερνήσεις κτλ. Και υπήρξε ένας κανονισμός ο οποίος θα εφαρμόζεται για περιορισμένο αριθμό προϊόντων θα αφορά το τελικό προϊόν προς τον καταναλωτή και θα, έχει, ε, θα υπάρξει ένα πιλωτικό σχέδιο πέντε ετών. Αυτά, ήτανε, αυτά είναι οι τρεις άξονες στους οποίους βασιστήκαμε. Ξέρουμε ότι ο πρωτοστατευτισμός δεν έχει να κάνει με αυτό το θέμα και ξέρουμε ότι οι διαθεσμικές ε, σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Επομένως, δεν θα πρέπει να ξαφνικά να μας λέτε ότι αποσύρετε μία πρόταση. Τα, αυτά τα πέντε χρόνια νομίζω ότι εμείς κάναμε τη δική μας δουλειά. Αλλά νομίζω ότι η Κομισιόν έχει πρόβλημα και κυρίως το Συμβούλιο δημιούργησε πρόβλημα, ε, το οποίο αρνείται να προχωρήσει και να κάνει κάτι ε, για κάτι που ζητάει ο επιχειρηματικός κόσμος. Ένα από τα λίγα πράγματα που αξίζουν τον κόπο. τον κόπο. Δημιουργήθηκε προσδοκία, δημιουργήθηκαν ε, ελπίδε. αλλά κάποιοι τώρα δεν θέλουν να αναλάβουν τι ευθύνε του. Φυσικά αυτή η δουλειά θα πρέπει να προετοιμαστεί με οργανώσει. και ξέρω ότι σε ορισμένε ε, χώρε έχουν ε, τεράστια προβλήματα αυτέ οι οργανώσει. Ξέρω ότι υπάρχουν κυβερνήσει που μπορούν και διμερώς να πάρουν μέτρα. Δεν λένε μονολόγια, κάνουν πράγματα, αλλά διμερώς. Φυσικά θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και στο εσωτερικό του ΠΟΕ. Αλλά νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής τουλάχιστον έδειξε την ικανότητά του να ακούει. Εδώ στην Ευρώπη κάνουμε ρυθμίσεις για τα πάντα, ακόμα και για την ενιαία χειραποσκευή όταν παίρνουμε το αεροπλάνο. Αλλά για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αγγίζει την καρδιά του επιχειρηματικού μας, του επιχειρηματικού μας κόσμου, τι δείχνουμε φόβο. Ευχαριστώ. Από τους πράσινους, ο κύριος Ζαντό για 2,5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Δεν διέφυγε της προσοχής σας ε, ότι διανύουμε μια σοβαρότατη κρίση και πολλοί συμπολίτες μας ε, αγωνιούν, ε, ανησυχούν για τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, τα έχουν λίγο χαμένα και ταυτόχρονα υπόκειται σε αντιφατικές πιέσεις. Από τη μία τους λέμε καταναλωτές καταναλώστε περισσότερο για να τονώσετε την οικονομία και να σώσετε τη θέση, τη απασχόλησης και να ενισχύσετε την, οικονομική, την οικονομική ανάπτυξη. Από την άλλη τους λέμε «Ε, καταναλώνετε υπερβολικά, με κακό τρόπο, ε, βυθίζουμε τον πλανήτη. Προσπαθούμε όμως ταυτόχρονα να δώσουμε κάποια εφόδια στον καταναλωτή για να αντιμετωπίσει την παγκοσμιοποίηση και να έχει κάποια όπλα να αντισταθεί. Και ταυτόχρονα του λέμε ότι πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην ε, παγκοσμιοποίηση και δεν θα πρέπει να δίδουμε στον προστατευτισμό. Τα ωφέλη του, της, της φιλελευθεροποίησης είναι προφανή. Δεν πρέπει να φοβάστε να ενισχύσετε τα δικαιώματα του καταναλωτή, εκτός κι αν δείχνει κρίση ότι τελικά αυτός ο φιλελευθερισμός έχει αποτύχει παταγωδός. Και δεν μπορείτε, εν αυτή περίπτωση, απλώς να μας προτείνετε μόνο να ενισχύετε τον έλεγχο τη εισαγωγή των προϊόντων, γιατί Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο όπου οι πολίτες πρέπει να είναι πρωταγωνιστές, πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής. Το Made in δεν είναι η θαυματουργή λύση, ούτε αν απαντά όλε τι ερωτήσει για το κοινωνικό ή το περιβαλλοντικό dumping. Είναι παρόλα αυτά ένα μηχανισμό σημαντικό, ένα σημείο αναφορά που επιτρέπει στον καταναλωτή να είναι ο πρωταγωνιστής τη ζωή του, να έχει δικαίωμα στη γνώση, στην επιλογή. Κύριε Επίτροπε, σα ζητούμε να φροντίσετε, να μεριμνήσετε για την ενίσχυση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να παραγωνίζει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει και το Συμβούλιο να αποφύγει ένα τέτοιο παραγωνισμό του Συμβουλίου. Πολύ σωστά επισημάναμε την απουσία του Συμβουλίου από τη συζήτηση, αλλά στην κρίση αυτής της παγκοσμιοποίησης ας μην περιμένουμε άλλο για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των συμπολιτών μας των καταναλωτών δηλαδή. Ευχαριστώ. ECR, η κυρία Γκέρλινγκ, για ένα λεπτό. Thank you. Ευχαριστώ. Είχα ανέκαθεν ε, ανησυχίε για την πρόταση κανονισμού. Μπορεί η υποχρεωτική ένδειξη προέλευση να αποφύγει ή να αποτρέψει την απομίμηση παραποίηση προϊόντων. Πόσο αποτελεσματική είναι στη, για την ιχνηλασιμότητα και την προέλευση των προϊόντων δεδομένη τη περιπλοκότητα τη αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων σε ένα παγκοσμιωμένο κόσμο. Το κόστο ε, μια ένδειξη προέλευση ε, είναι μήπω υπερβολικό. Όλε αυτέ οι ερωτήσει είναι εύστοχε και εύλογε. Πέραν όμω των εμπορικών ρυθμίσεων και τη συμβατότητα με τι διατάξει του ΠΟΕ, αναγνωρίζω, αντιλαμβάνομαι το αίτημα του καταναλωτή να γνωρίσει την προέλευση των προϊόντων που καταναλώνει για πολλού και διάφορου λόγου. Για παράδειγμα, θέλουν να στηρίξουν την εθνική του βιομηχανία, το δικαίωμα επιλογή με εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την προέλευση των προϊόντων. Οπότε, λέω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι και εκείνη η ώρα να προχωρήσουμε. Ε, να μπορώ, μπορώ πια να μπω σε ένα κατάστημα, να ε, στρέψω το κινητό μου Προ ένα προϊόν και να μάθω από πού προέρχεται αυτό το προϊόν. Αυτή είναι η ελευθερία που μας δίνει και η δυνατότητα που μας δίνει η νέα τεχνολογία. Δεν είναι προστατευτισμός. Ας δώσουμε στους καταναλωτές πληροφορίες που απαιτούν. Είναι σημαντικό το θέμα. Μην παρατηθείτε λοιπόν από την προσπάθεια αυτή. Η αυτή. Ο κ. Σαλβίνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Στρέφουμε εδώ και στους ακροατές μας στο ίντερνετ. 112 εργάτες χθες πέθαναν στο Μπαγκλαντές, μεταξύ των οποίων γυναίκα και παιδιά. Ε, κατασκεύαζαν με ένα δολάριο τη μέρα ε, κα, ε, κλωστοφαντουργικά τα οποία πολλούνται στην ε, Ευρώπη. Τι κάνουμε για αυτούς ένα λεπτού, ενός λεπτού σιγή. Το θέμα είναι τι καταναλώνουμε, τι φοράμε. Δεν ξέρω αν αυτό που φοράω ε, παράχθηκε στο, στη χώρα μου, στην Ιταλία ή κάπου στο Μπαγκλαντές. Εγώ θα ήθελα να το ξέρω. Θα ήθελα να το ξέρω. Και εγώ και τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται. Υπάρχουν οι πολυεθνικές. Ε, υπάρχουν ε, τα παπούτσια του Πακιστάν, υπάρχουν τα οποροκυπευτικά από το Μαρόκο. Κανένας δεν ενδιαφέρεται αν χρεοκοπούν χιλιάδες επιχειρήσεις εδώ, αν χάνονται θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Αλλά αν χάνονται εδώ σημαίνει ότι ίσως κάπου αλλού, ε, στην άλλη άκρη του κόσμου, ε, προσλαμβάνουμε ένα παιδί και το πληρώνουμε ένα δολάριο τη μέρα. Επομένως, ε, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Βραζιλία, το Μεξικό και η Ιαπωνία που βάζουν το σήμα ενημερώνουν τους καταναλωτές για το πού φτιάχνουν τα προϊόντα τους. Εμείς όμως δεν ενδιαφερόμαστε, δεν μας νοιάζει. Και σα εκπλήσει που οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν καταλαβαίνουν την Ευρώπη και είναι μακριά, αισθάνονται μακριά. Ε, όμως οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για τα εργοστάσια στη Λομβαρδία που, που κλείνουν. Αυτή η Ευρώπη όμως ε, είναι τραγική. Ας μας σώσει ο Θεός από αυτή την Ευρώπη. Από την ΚΟΕ, ο κύριος Σκόλτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπή, η ομάδα μου συμμερίζεται τη στεναρή κριτική του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αδικαιολόγητη παρελκυστική ε, τακτική ε, του Συμβουλίου. Έχω δικαίωμα οι καταναλωτέ να γνωρίζουν την προέλευση ενό προϊόντο. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αμελητή να καταθέσει νέα νομοθετική πρόταση και να υιοθετήσει την ηλυμένη απόφαση ε, του Κοινοβουλίου ακριβώς επειδή αρνείται το Συμβούλιο. Οι πολίτε θέλουν να μαθαίνουν περισσότερα από το όνομα μιας χώρας που μπορεί να είναι μόνο το πρώτο βήμα. Τον 21ο αιώνα είναι σημαντικό για τους καταναλωτέ στην παγκοσμιοποίηση να γνωρίζουν τι γίνεται στην παραγωγή, ανεξάρτητα από τη χώρα. Να τηρούνται τα κοινωνικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα προϊόντα να μην βλάπτουν την υγεία τους και να μην βλάπτουν και το περιβάλλον και το κλίμα. Αυτό είναι το fair made, το fair trade και η διαφάνεια για τους πολίτες. Και καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγωνιστεί και στον ΠΟΕ για εξυγχρονισμό των κανόνων του παγκοσμίου εμπορίου και όχι να κρυβόμαστε πίσω από τους ισχύοντες κανόνες θα πρέπει το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ παγκοσμίω να στιγματιστούν για να μην πέσουμε θύμα της παγκοσμιοποίησης και των αλυσίδων παραγωγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φιέλνερ. λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω το γεγονός ότι η Κομισιόν έχει αποσύρει αυτόν τον καονισμό. Χθε συζητούσαμε τα σήματα καταγωγής και είδαμε πόσο περίπλοκοι μπορεί να είναι αυτοί οι κανόνες. Μας ανησυχεί το γεγονός από το ότι μονομερός η Ευρωπαϊκή Ένωση επρόκειτο να εισάγει τέτοιους κανόνες. Ε, για το πουκάμισό μου, ας πούμε, το, το βαμβάκι από πού προέρχεται, από την Ιταλία. Ε, το επεξεργάστηκαν σε εργοστάσια στην Ιταλία, μετά πήγε στο Χονγκ Κόνγκ για μια άλλη επεξεργασία και ήρθε στη χώρα μου. Υπάρχουν πολύ, πολύ διαφορετικές συνθήκες από εργοστάσιο σε εργοστάσιο σε διαφορετικές χώρες. Εμείς μιλάμε για υποχρεωτική ένδειξη ε, της καταγωγής προϊόντων στην, που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είχαμε σκεφτεί αυτό, αλλά τελικά αποφασίσαμε να το κάνουμε γιατί ήταν πολύ ακριβό για τους, κατα... για τους παραγωγούς μας. Γιατί τώρα να το επιβάλλουμε αυτό για τα εισαγόμενα είδη. Ε, δεν ξέρω, οι καταναλωτές το θέλουν αυτό. Αν το ήθελαν οι βιομήχανοι θα χρησιμοποιούσαν από μόνοι τους αυτό το made in χωρίς να τους αναγκάσουμε εμείς. Ας, ας το αφήσουμε να πεθάνει από μόνο του, εάν δεν το θέλουν οι βιομηχανοί και οι κατασκευαστές αυτό το σήμα. Μία μπλε κάρτα, τη δέχεστε? Με το, με, ανάμεσα σε μένα και στον κύριο Φιέλνερ έχουμε συνέχεια μπλε κάρτες. Τελικά κύριε Φιέλνερ, δηλαδή μόνο τα εύκολα θέλετε να κάνουμε. Επειδή είναι δύσκολο να ξέρουμε ποια είναι η καταγωγή ενός προϊόντος, το οποίο το υλικό έρχεται από μια χώρα, ε, το επεξεργαζόμαστε σε άλλη χώρα και, το, και η τελική επεξεργασία γίνεται σε μια τρίτη χώρα, δεν πρέπει να λέμε τίποτα. Δηλαδή εμεί θα κάνουμε τα εύκολα μόνο. Τα περίπλοκα τα ξεχνάμε. Γιατί είμαστε εδώ πέρα. Για να κάνουμε τα εύκολα, τα απλά. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε ε, στον καταναλωτή από πού έρχεται ένα προϊόν. Δεν θα πρέπει να βάζουμε κανένα σήμα το οποίο θα λέει την προέλευση ή καταγωγή του προϊόντος αυτού. Καλό αυτό, ε. Εύκολο είναι. Δεν θα είναι πιο σωστό, κύριε Φιέλντε, να πείτε ότι εσεί για... προσπίζεστε τα συμφέροντα, α πούμε, τη χώρα σα ή των εταιριών σα, εν Ή επίση, επειδή αδιαφορείτε εντελώ για την πραγματικότητα τη βιομηχανία, α πούμε, γι' αυτό έχετε αυτή τη θέση. Δεν θα είναι πιο σωστό και τίμιο να το πείτε αυτό. Ευχαριστώ. Πραγματικά γίνεται παράδοση μεταξύ μας. Αντίθετα όμως πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει και στα δύσκολα. Και αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε, αν έχουμε περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερο προστατευτισμό, περισσότερα τελωνια... περισσότερους τελωνιακούς δασμούς, τότε δεν νομίζω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί τελικά ε, και ούτε πρόκειται να φτιάξουμε περισσότερα μπλουζάκια, ας πούμε, σε σχέση με το Βιετνάμ. Άνθρωποι στο, Βιετνα... στο Βιετνάμ μας είπαν ότι δεν θα μπορούσαν να ζήσουν αν δεν τους επιτρέπουμε να συνεχίσουν τις κλωστοϊφαντουργικές τους ε, δραστηριότητες μόνος με φτιάχνοντας παπούτσια. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε καλά. Λάγκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Γιατί είμαστε κατά της πρότασης, ε, στα αλήθεια. Ένα, ένας είναι ο λόγος. με μονομένη παραγωγή και με μονομένη έμποροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν το συμφέρον να μην ξεκαθαρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα τους. Αγοράζουν φτηνά παγκοσμίω και πουλούν ακριβά στην Ευρώπη με την επίφαση ότι έχουν παραχθεί σε λογικές συνθήκες τα προϊόντα στην Ευρώπη. Αυτά είναι συμφέροντα μεμονωμένα οικονομικά ορισμένων παραγωγών και ορισμένων εμπόρων και δεν θα πρέπει να ενδώσουμε. Ε, χρειαζόμαστε διαφάνεια στην αλυσίδα της προμήθειας. Θα πρέπει ο καθένας να γνωρίζει την προέλευση και να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στην Ένωση. Γι' αυτό εμένα με ενδιαφέρουν τα εξή δύο ερωτήματα. Πρώτον, τι, τι τρέχει στο Συμβούλιο. Θέλει επιτέλους το Συμβούλιο από κοινού να προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον κοινωτικό πνεύμα και ε, στο συμφέρον των καταναλωτών ή ενδίδει σε οικονομικά συμφέροντα μεμονωμένα και ιδιωτελή και απεμπολεί την ευρωπαϊκή μέθοδο γιατί φοβούμαι ότι αυτό τον καιρό, μάλλον το δεύτερο υπερισχύει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν ενδιαφέρεται να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά να προασπίσει ιδιωτελή εμπορικά οικονομικά συμφέροντα. Δεν επιτρέπεται αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Ερώτηση δεύτερη προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσεί με το πλευρό ποιανού είστε, είστε στο πλευρό του Συμβουλίου με τα ε, οικονομικά ιδιωτελή συμφέροντα ή ε, στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλει να μεταξελίξει την Ένωση με την κοινοτική μέθοδο. Ονορεύολε Μάντερς. λεπτό. γίνεται τώρα για τα θεσμικά προβλήματα, προβλήματα με τον ΠΟΕ. Στην Ευρώπη εμείς νομοθετούμε για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης και την τονίζουμε. Ε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε ε, την ανθρωπιά στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και καλά κάνουμε. Και κάνουμε και νομοθεσία για το περιβάλλον. <clears throat> Έχουμε τώρα προβλήματα. Εγώ είμαι δικηγόρος, ε, στο παρελθόν ήταν και ο Επίτροπος και νομίζω ότι θα πρέπει να επιλέξετε άλλη οδό. Δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η σήμανση προέλευση στα προϊόντα τα εισαγόμενα. Να το αντιστρέψουμε, να πούμε να είναι θελούσια ε, η σήμανση. Made in EU, made in Germany. Αλλά να γνωρίζουν όλοι τι ισχύει ε, σε μια χώρα και ότι θα πρέπει να ε, παράγονται όλα τα στοιχεία του προϊόντος στη χώρα αυτή, να είναι εθελούσια, αλλά όχι ε, αυθαίρετη ε, η σήμανση. Να λέμε ένα προϊόν έχει φτιαχτεί η Γερμανία στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να λέει το κουστούμι made in Germany και να έχουν ράψει μόνο τα κουμπιά και όλα τα άλλα να τα έχουν κάνει σε χώρες φθηνής παραγωγής αλλού. Γιατί βασικά κινέζικο κουστούμι φοράω, ακόμα και να έχουν ραφτεί τα κουμπιά στη Γερμανία. Ευχαριστώ. La ehm, Ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ. Οι καταναλωτέ θέλουν να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα τρόφιμα. Είναι σωστό λοιπόν που εξετάζουμε σήμερα του κανόνε προέλευση. Βέβαια, αυτό που οι καταναλωτέ επιθυμούν να μάθουν είναι η χώρα, τη χώρα καταγωγής θέλουν να βλέπουν το Made in England, Made in France, ε, στη Γαλλία, στην Ιταλία, κατασκευασμένο στην ε, Γερμανία και ούτω καθεξής. Μάλιστα, λίγοι καταναλωτές μπορεί να θέλουν ε, να βλέπουν Made in στη Ρουμανία. Θέλουν, δεν θέλουν βέβαια να βλέπουν απλώς φτιαγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω μία ελπίδα στο κεφρούδα ότι οι κανόνε αυτοί δεν θα είναι ένας ακόμη μηχανισμό για να μας βάλουν και πάλι στο δρόμο του ευρωπαϊκού υπερκράτους. Ο κύριος Προύστ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω μείνει εμβρόντιτος και βαθύτατα ανήσυχος για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσύρει τον κανονισμό, την πρόταση κανονισμού Made in για την ένδειξη προέλευσης με πάνω από 85% ε, ψήφους υπέρ με τη σχετική πρόταση πριν από δύο χρόνια. Και παρόλα αυτά περιφρονείται τη γνώμη των ε, Ευρωβουλευτών και άρα και των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Μάλιστα το Made in αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της ενημέρωσης ε, προς τον καταναλωτή και είναι πολύ αρνητικό το μήνυμα δεδομένης της δυσπιστίας που υπάρχει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κοινωτικά θεσμικά όργανα εκ μέρους των πολιτών. Λέτε ότι ο βασικός λόγος της μελλοντικής απόσυρσης είναι ότι έχει πλέον απερχιωθεί μετά την ομολογία του ΠΟΑ για το cool case ε, η σχετική νομοθεσία. Σταματήστε να μας αντιμετωπίσετε σαν να είμαστε αφελείς θα υποβάλει νέα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ομολογία του ΠΟΕ. Πώ εξηγείτε ότι η Βραζιλία, ο Καναδά και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν βρει τρόπο να συμφιλειώσουν την νομοθεσία του για το Made in και το σεβασμό των υποχρεώσεών του προ τον ΠΟΕ. Μήπω θέλετε να αποσύρετε τον κανονισμό για να σώσετε τα προσχήματα όταν βλέπετε την ανικανότητα του Συμβουλίου να καταλήξει συμφωνία. Δυστυχώ βρίσκεται σε ύφεση η ανταγωνιστικότητά μα ε, το MADE είναι ένας μηχανισμός που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, είναι παράλογο να το καταργούμε. Σας εύχομαι πραγματικά το 2003 να βρείτε μια πιο λογική διέξοδο για το θέμα αυτό και ελπίζω επιτέλους ε, το Συμβούλιο να ξυπνήσει. Η κυρία Μπαντία, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε σε αυτή τη φάση της συζήτησης ήδη έχουν ε, παρουσιαστεί όλα τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της διατήρησης του κανονισμού. Είχαμε τη συζήτηση για την ενημέρωση για την προέλευση, για τους κανόνες προέλευσης. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και πολύ σημαντικό επίσης είναι το θέμα της διαφάνειας. Εγώ θα ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητα που έχει το θέμα αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε και το λέμε καθημερινά σε εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων με το μισό τζίρο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, έχουν δημιουργήσει το 80% των θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε, είναι καθήκον μας να μεριμνήσουμε ώστε οι επιχειρήσεις αυτές που εμπλουτίζουν την οικονομία και δημιουργούν θέσεις εργασίας να δραστηριοποιούνται σε συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού απέναντι στα εισαγόμενα προϊόντα. Ξανασκεφτείτε λοιπόν κύριε Επίτροπε την πρόταση για απόσυρση του κανονισμού. Γιατί με τέτοια απόσυρση ουσιαστικά θα αφήσουμε ανήμπορε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει μα. Δεν θα συμβάλλουμε ούτε στην οικονομική ανάπτυξη ούτε στη δημιουργία απασχόληση. Θέλουμε τον κανονισμό αυτό γιατί οι καταναλωτέ μα έχουν την ικανότητα και θέλουν να γνωρίζουν τι καταναλώνουν, την προέλευση των προϊόντων και θέλουμε οι κοινωνικέ προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρούνται και να διαφυλάσσονται όχι μόνο εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στι τρίτε χώρε. Παρακαλώ λοιπόν, ξανασκεφτείτε την πρότασή σα για απόσυρση του κανονισμού. Αν θέλετε να τον αναθεωρήσετε, αναθεωρήστε τον, αλλά μην τον παραμερίζετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κούτα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτός ο κανονισμός που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 από το Κοινοβούλιο είναι η σωστή απάντηση στο αίτημα βελτίωσης της διαφάνειας και της πληροφορίας των καταναλωτών στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα που εμφανίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτός ο κανονισμός είναι χρήσιμος γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σωστή νομοθεσία ε, σε αυτόν τον τομέα. Είναι κρίμα λοιπόν που η Κομισιόν αποφάσισε να αποσύρει αυτόν τον κανονισμό και να αγνοήσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών να γνωρίζουν την προέλευση προϊόντων, να ξέρουν αν τηρούνται οι κανόνες ε, για το περιβάλλον και την ασφάλεια. Ε, περισσότερες πληροφορίες και περισσότερη διαφάνεια για τους καταναλωτές δεν σημαίνει μεγαλύτερος προστατευτισμός. Αυτό θα να σας πω κύριε Επίτροπε. Τόια ένα λεπτό. Η πρόταση απόσυρσης του καονισμού ήταν σαν κεραυνός σε Ε, δεν είναι καλό σημάδι, κύριε Επίτροπε, στις διαθεσμικές σχέσεις μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Ξέρετε πολύ, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το κάνετε. Κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, πίσω από τα στοιχεία του ΠΟΕ. Από τα λόγια σας όμως προκύπτει, ότι δεν είσαστε πεπισμένος για αυτόν τον καονισμό ότι θα είναι δαπανηρό, ότι είναι προστατευτικό, προάγει τον προστατευτισμό κτλ. Όλα αυτά δεν είναι πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι είσαστε ανίκανοι ω Κομισιόν να είσαστε συνεπείς ε, και να προχωρήσετε προ αυτόν τον δρόμο. Ακούσατε Ακούσατε τι είπαν οι ευρωβουλευτέ από όλο το πολιτικό φάσμα, ακόμα και οι ευρωσκεπτικιστές. Ε, αν μετά από αυτά που ακούσατε, εσείς θα, είσαστε τόσο θα συνεχίσετε να είσαστε τόσο σκεπτικιστές και να υπερασπίζεστε κάποια λίγα ιδιωτικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των καταναλωτών, δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Ονορεύολε δύο λεπτά. Ο Επίτροπες μα είπε ότι δεν υπάρχουν προοπτικέ συμβιβασμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ποιο το είπε αυτό κύριε Επίτροπε, Ποιο προσπάθησε να βρει μια μέση λύση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων που, που να συναντηθούν και να βρεθεί ένα συμβιβασμό. Είπατε ότι δεν εφαρμόζεται στα εσωτερικά εγχώρια προϊόντα. Φυσικά. Φυσικά, προφανώς. Εμείς πρέπει Πιστεύουμε ότι πρέπει να σταματήσετε, να μην προχωρήσετε με την απόσυρση αυτή, να αναλύσετε τι κάνανε οι άλλες χώρες που έχουν παρόμοιο κανονισμό και μέσα από αυτή την ανάλυση να μας παρουσιάσετε ενδεχόμενες τροποποιήσεις στην πρόταση που ήδη έχουμε ψηφίσει. Αν είσαστε πεπισμένος ότι αυτή η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στον σημερινό και δεν σέβεται το σημερινό μηχανισμό του ΠΟΕ, τότε να μας προτείνετε αλλαγές. Αλλά δεν μπορούμε στο εσωτερικό του ΠΟΕ να είμαστε χώρες που θα έχουμε κάποιον κανονισμό και χώρες που δεν θα έχουν τέτοιον κανονισμό. Δεν είναι σωστό αυτό. Θα έχουμε διαφορετικούς δηλαδή κανόνες ανταγωνισμού και αυτοί οι κανόνες κάποιους τιμωρούν και κάποιους όχι. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να πει τη γνώμη του πριν αποφασίσει η Κομισιόν να προχωρήσει στην απόσυρση αυτή. Τέλος πάντων, εμείς σημειώνουμε τη δήλωσή σας Θέλουμε να πιστέψουμε ότι ξέρετε τι κάνετε. Εμείς σήμερα διατρανώνουμε τη θέση μας. Και θα το πούμε και με ψήφο πολύ ξεκάθαρη. Σας ζητούμε λοιπόν να σταματήσετε και να μην προβείτε σε αυτή την απόσυρση, να ακούσετε τη γνώμη του Κοινοβουλίου, να δεσμευτείτε ότι θα επαναφέρετε το διαθεσμικό διάλογο και θα προβλέψετε να γίνει μια συνάντηση αρχικά άτυπη με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα για να αξιολογήσετε την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησεων και εξέβρεσης λύσεων που θα συμμεριζόμαστε όλοι, ούτω ώστε να βρεθεί ένα συμβιβασμό, ε, κύριε Επίτροπε. Γιατί εσεί εκπροσωπείτε την Ευρώπη και θα πρέπει να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα τη Ευρώπη. Ο κύριο Ταραμπέλα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε έδωσα μάχη προκειμένου μέσω κατάλληλη σήμανση να έχει ο καταναλωτή πρόσβαση σε σωστή ενημέρωση. Και ε, θέση της, ε, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εξασφαλίσει τα μέσα στον πολίτη για να ενημερώνεται. Η ένδειξη προέλευση εντάσσεται σε αυτή την προοπτική και μάλιστα πολλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ αυτής της πρότασης ε, καθώς και της ενα... θέσπισης εναρμονισμένων κυρώσεων σε περίπτωση παράβαση. Δυστυχώ κολλήσει το Συμβούλιο μπλοκάροντας την νομοθετική διαδικασία. Τώρα όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρί καμία συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλει να αποσύρει τον κανονισμό. Ενορχιστρωμένοι λοιπόν από τα θεσμικά όργανα, έχουμε μία ε, ήττα τη προάσπιση του δικαιώματο του καταναλωτή, που δεν συνάδει, δεν είναι συμβατή με το εμπόριο, αν είναι δυνατόν. Ε, άλλωστε το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να τονώσει την ε, παραγωγή αλλά και την απασχόληση στις ε, ευρωπαϊκές επιχείρησεις. Για μια ακόμη φορά οι εταιρείε που ασχολείται με την ε, παρασκευή των προϊόντων δεν αναδεικνύονται και δεν προωθούνται. Ευχαριστώ. Πάμε στο Catch the Eye. Έχουμε 10 αιτήματα για ένα λεπτό καθένας. Ο πρώτος ομιλητής παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, με εκπλήσει η τακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πρώτη ανάγνωση. Το Κοινοβούλιο διατράνωσε τη θέση του. Παρόλα αυτά, τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν. Αλλά είναι πραγματικά περίεργη η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν το άλλαξαν, ε, δεν το το άλλαξαν για τον ΠΟΕ. Αυτά που μας λέτε και σήμερα είναι τελείως απαραδεκτά. Αντί να εργαστείτε για να βρείτε μια λύση συμβατή με τον ΠΟΕ, είδατε πλούστατα την πρόταση. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα εγγυηθείτε αυτό που έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο, οι εισαγωγέ από τις τρίτε χώρες να είναι αντίστοιχε με τη δική μας παραγωγή και στα κοινωνικά και στα περιβαλλοντικά και στα εργατικά ε, δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον σκοπεύει πριν αποσύρει νομοθετική πρόταση να ενημερώνει για να μην μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το Κοινοβούλιο στις αποφάσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλβέστρης. Το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με 529 ψήφους τον κανονισμό για την υποχρεωτική ε, αναγραφή της καταγωγής. Ε, είναι ευρύτατη η πλειοψηφία, κύριε Επίτροπε. Δεν θα έπρεπε να αποσύρετε τον κανονισμό. Είναι σημαντικό αυτό το σήμα για κάποια προϊόντα. Παραδείγματο χάρη στην Πούλια, στην Καλαβρία, στο νότο της Ιταλίας, στη Βασιλικάτα, στην Πολύζε. Ε, έχουμε ε, κατακλειστεί από κινέζικα προϊόντα και χιλιάδες μικρές ε, εταιρείε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κλείσει, δημιουργώντας χιλιάδες ανέργους. τα παιδιά τα οποία δουλεύουν σε εταιρείε στην Κίνα παράγουν ευθυνά προϊόντα και αυτό κοστίζει σε εμάς. Επιπλέον, σε αυτό το κόστος προστίθεται και το κοινωνικό κόστος. Ε, η εκμετάλλευση των παιδιών, καμία προστασία για το περιβάλλον, για τους ανήλικους, ε, για τις ε, εγγύους γυναίκες. Όλοι, ακόμα και εσείς κύριε Επίτροπε, στην Ευρώπη ξέρουμε γιατί τα κλωστοφαντουργικά προϊόντα ή τα προϊόντα υποδηματοποίησης των τρίτων χωρών είναι τόσο ανταγωνιστικά, τόσο φθηνά. Γιατί αντιμετωπίζονται οι, εργαζόμενοι ως σκλάβοι. Δεν θα έπρεπε λοιπόν ο καταναλωτή να ξέρει ε, από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Με το να αποσύρετε την πρόταση αυτού του κανονισμού, κύριε Επίτροπε, ε, τελικά ποια συμφέροντα ε, εξυπηρετείτε. Τα, τα συμφέροντα των εταιριών που παράγουν νόμιμα, των μικρών ας πούμε επιχειρήσεων που παράγουν παπούτσια στην Ευρώπη ή των πολυεθνικών ας πούμε που μεθεγκατίστανται τις εταιρείες που πληρώνουν ένα τίμιο μισθό στις, ε, στην Ευρώπη ή αυτό που εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους και τους αντιμετωπίζουν σαν σκλάβους. Σας παρακαλώ, ε, προσπαθήστε να κάνετε κάτι για να κερδίσει και εσείς και η Ευρώπη αξιοπιστία. Ο κύριος Δανέλης. Κύριε Επίτροπε, θα αναφερθώ στα ιδιαίτερα προβλήματα της εμπορίας εμπορευμάτων όπως τα νοπά γεωργικά προϊόντα μπορεί ένα γεωργικό προϊόν που εισάγεται από τρίτες χώρες όπου το κόστος παραγωγής είναι σαφώς χαμηλότερο να προωθείται στην αγορά της ευρωπαϊκής ένωσης ως ευρωπαϊκό από τη στιγμή που υποστεί μεταποίηση σε κράτος μέλος της ένωσης ακόμη και αν αυτή η μεταποίηση δεν αλλάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή την ειδική υφή <clears throat> του πρωτογενούς προϊόντος. έτσι οδηγούμαστε εύκολα σε παραπληροφόρηση του καταναλωτή ο οποίος μπορεί να διαβάζει στην ετικέτα του προϊόντος ότι η επιλογή του είναι προϊόν της Ένωσης και να αγνοεί ότι η πρωτογενής ύλη παράχθηκε σε χώρα εκτός της Ένωσης. Η προστασία του καταναλωτή και η διασφάλιση του θεμητού ανταγωνισμού δεν συνιστούν προστατευτισμό, αλλά υποχρέωση της Ένωσης. Ευχαριστώ. Kadenbach. Κύριε κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σήμερα ε, αισθάνομαι τριπλή εγκατάλειψη. Πρώτον, με έχει εγκαταλείψει το Συμβούλιο, που ως εταίρος μας λείπει πάρα πολύ σήμερα. Αλλά διπλά μας έχετε εγκαταλείψει εσείς και εμένα ως βουλευτή και ως καταναλώτρια. Γιατί καταναλωτές 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους έχουμε και το συμφέρον τους είναι να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Ε, και τα χρησιμοποιούν αυτά τα εμπορεύματα. Σε όλα τα ευρωβαρόμετρα το βλέπουμε. Οι καταναλωτέ θέλουν να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Δεύτερον, αισθάνομαι ότι με έχετε εγκαταλείψει κι εσεί ε, ω βουλευτή κύριε Επίτροπε. Πριν από δύο χρόνια το κοινοβούλιο μα ε, έλαβε ξεκάθαρη θέση. Και εσεί μαζί με το Συμβούλιο είχατε την ευκαιρία τη θέση αυτή να τη διαπραγματευτείτε. Ε, τώρα είναι φτηνό επιχείρημα, μας λέτε δεν το επιτρέπει ο ΠΟΕ διαπραγματευτικός εταίρος είναι και ο ΠΟΕ. Έχετε και τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να διαπραγματεύεστε από κοινού και να αλλάζετε αυτά που αποφασίζουμε εμείς ε, να τα προσαρμόζετε. Η απειλή σας η σημερινή μάλλον ήταν για να μας ξυπνήσει και ελπίζω να μην είναι πραγματικότητα. Περιμένω θέσεις διαπραγμάτευσης που να συνάδουν και με τον ΠΟΕ αλλά και με τις προσδοκίες των Ευρωπαίων. Φερέιρα. Ευχαριστώ. Η τροπή της κατάστασης δείχνει για μια ακόμη φορά την πραγματική θέση και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο πλευρό αυτών που είναι κατά τη αναφορά σε ένδειξη προέλευση. Προασπίζει αυτού που επωφελούνται από την απορρίθμιση και τη φιλελευθερωποίηση του παγκοσμίου εμπορίου, δηλαδή τι πολυεθνικέ μεγάλου εισαγωγή και δια... του μεγάλου διανομή. Τάσετε υπέρ τη ελεύθερη επιλογή και τη διαφάνεια για του καταναλωτέ. Αυτά τα αφήνει κατά μέρο δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί ε, ταχθήκαμε υπέρ τη ένδειξη ε, προέλευση των προϊόντων. Θεωρούμε ότι είναι ένα μηχανισμό για να προστατεύσουμε και τι επιχειρήσει ε, τη Ευρώπη, να πατάξουμε το κοινωνικό και περιβαλλοντικό dumping. Είναι ένα μηχανισμό που ούτω ή άλλω δεν τροποποιεί άρδιν τι οικονομικέ και εμπορικέ πολιτικέ. Είναι πολύ περίπλοκη μερικές φορές ε, γεωγραφικά η αλυσίδα τώρα της διανομή, η αλυσίδα της διανομής. Θα πρέπει να αντιταχθούμε στο προστατευτισμό των μεγάλων συμφερόντων ε, εις βάρος ε, του γενικού συμφέροντος, του συμφέροντος των εργαζομένων και των, επιχειρήσεων της Ευρωπαϊ... των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Μοργάντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται να προστατεύσει τους ε, πολίτες. Η φωνή τους δεν μετράει. Ε, το Κοινοβούλιο όμως ε, εκπροσωπεί αυτούς τους πολίτες και εκφραστήκαμε ως Κοινοβούλιο ακριβώς επί του θέματος αυτού. Αυτός ο κανονισμός μας εξυπηρετεί. Θα μας δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και θα γνωρίζουν οι καταναλωτές, θα αγνοούν και δεν θα αγοράζουν τα, τις απομιμήσεις και τις μαϊμούδες με τις οποίες κατακλείζονται οι αγορές μας. Ε, δεν σας ενδιαφέρει προφανώς ε, να επειρασπιστείτε την ε, βιομηχανία που για μας είναι πολύ σημαντική. Ας συζητήσουμε για τα τελωνία. γιατί τα θέματα βιομηχανίας και τελωνία είναι πολύ συνδέονται. Ελπίζω ότι όλη η δουλειά που έχει γίνει να μην πάει χαμένη. Ελπίζω να βρούμε μία συμφωνία και με το ΠΟΕ. Σας πιέζει να κινηθείτε προς αυτήν την κατεύθυνση και δεν μπορεί να παραμείνετε κουφοί απέναντι στις εκκλήσεις μας. Δεν μπορεί να κοφεύετε απέναντι στις εκκλήσεις του λαού και των πολιτών. Οι δηλώσεις του Επιτρόπου για την απόσυρση αυτής της πρότασης δημιουργούν αμφιβολίες για την ε, νομιμότητα αυτής της κίνησης. Αλλά επιπλέον δημιουργούν και τα εξή δύο προβλήματα. Καταρχάς αυτή η όπισθεν που κάνετε προστίθεται στην ε, σιωπή του Συμβουλίου που επί χρόνια συνεχίζεται. Ποιο είναι ο ρόλο τελικά του Κοινοβουλίου στην ε, διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Μα απογυμνώνεται, μα μειώνεται. Δεν σέβεστε την απόφασή μας και απλώς προάγεται έτσι η γραφειοκρατία σας. Αγνοείτε τη φωνή των πολιτών που εμείς ε, δημοκρατικά εκπροσωπούμε. Επίσης δεν υπάρχει ένα νομοθέτημα συνεπές ούτως ώστε να μην επιτρέψουμε τις αγορές μας να κατακλείζονται από φθηνά προϊόντα τρίτων χωρών. Αυτό είναι προζημίαν των καταναλωτών που μπορούμε ε, να τους εξαπατήσουμε για την ποιότητα των ε, προϊόντων που αγοράζουν. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς ένα πιο αποτελεσματικό έλεγχο και αυτός ο κανονισμός θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το να το ξεχάσετε σημαίνει ότι πετάτε το γάντι ότι δεν δίνετε αυτή τη μάχη. Ποια είναι η θέση σας, Κομισιόν. Θα ήθελα να επιτρέψετε η νομοθετική αυτή διαδικασία να συνεχίσει την πορεία της και να μην εμποδίσετε τον διάλογο ανάμεσα στους συνομοθέτες. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος, ε, κύριος Δεχούχτ. Uh, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση αυτή. Πολύ ζωντανή, οφείλω να ομολογήσω, τέτοια ώρα πρωί-πρωί. Πολλές ερωτήσεις έγιναν καταρχάς για τον ΠΟΕ. Οι αποφάσεις του ΠΟΕ είναι σαφείς, ξέρετε. Υπάρχουν ε, διευκρινήσεις για τους κανόνες που διέπουν τη σήμανση ως προς την προέλευση και ε, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρόταση του 2005 είναι πεπαλαιωμένη, ξεπερασμένη, γιατί έχει διαφορετική μεταχείριση στα εισαγόμενα και τα χώρια προϊόντα. Ας πούμε, είναι υποχρεωτική η σήμανση της προέλευσης μόνο για τα εισαγόμενα προϊόντα και μόλις τον Οκτώβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε για τις προϋποθέσεις αυτές και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τι λέγει λοιπόν το αρμόδιο όργανο του ΠΟΕ, έτσι ε, συντομία. Ε, τι... Ότι θα πρέπει ε, να ε, συνάδουν όλα αυτά με τη συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Ε, αυτό είπε η Επιτροπή Προσφυγών. Και θα πρέπει μεταξύ άλλων να συνάδουμε την ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους και διάφορες αντίστοιχες εμπορικές συμφωνίες, ιδιαίτερα προϊόντα εισαγόμενα δεν θα πρέπει να υφίστανται μειονεκτική μεταχείριση σε σχέση με τα εγχώρια. Γι' αυτό η πρόσφατη ε, νομολογία ε, έχει ε, ορίσει αντίστοιχα τη σήμανση των εθνικών προϊόντων, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να δικαιολογηθούν με βάση τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο. Έγιναν εδώ ορισμένα σχόλια που λέγουν, καλά, και με τις υπόλοιπε χώρες τι γίνεται. Δεν το δέχομαι αυτό το επιχείρημα γιατί τα όσα συζητούμε και αποφασίζουμε στον ΠΟΕ και σε όλες τις διαπραγματεύσεις είτε είναι ε, διμερείς είτε είναι πολυμερείς ε, θέτουν μεγάλη έμφαση στα τεχνικά εμπόδια ε, του εμπορίου και πώς αυτά θα έρθουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό από τους δασμούς για όριμες οικονομίες σαν τη δική μας. Δηλαδή δεν μπορούμε από τη μια να υψώνουμε διάφορα τεχνικά εμπόδια και τέτοια και να τα καταργούμε, αλλά όταν πρόκειται για την ετικέτα προέλευσης ε, κάνουμε τα στραβά μάτια. Ε, ορισμένοι άλλοι χρησιμοποιούν ένα επιχείρημα που λέει ότι αν ορισμένοι συμπεριφέρονται λάθος, γιατί να μην συμπεριφερόμαστε κι εμείς. Μα αυτό δεν είναι τρόπος λειτουργίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα βασικό εταίρο του ΠΟΕ. Ο Κόμις Ντάρθμουθ έκανε ένα ενδιαφέρον σχόλιο. Να γράφουμε Made in Germany. Α, έφυγε κιόλα. Ε, να αναφέρουμε τη χώρα Ιταλία, αλλά μα, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε κανόνες προέλευσης, έχουμε εσωτερική αγορά. Ε, τότε θα είχαμε πρόβλημα αν ήταν υποχρεωτικό αυτό, θα ήταν και αντίθετο με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Κύριε Ζαντό, δεν υπάρχει πια Made in France, είναι Made in European Union. Και κατά τα άλλα, τι θα κάνουμε τώρα. Ένα είδος άτυπων κανόνων για την προέλευση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με το αν μεγαλύτερο τμήμα του ε, προϊόντος έχει κατασκευαστεί στην Πορτογαλία ή στην Ιταλία. Μα ποτέ δεν πρόκειται αυτό να εφαρμοστεί. Το πολύ πολύ να πούμε made in Europe και αν θέλει κάποιος να προσθέτει κάτι άλλο ε, για να υπάρχει η επισήμανση του λόγω κράτους μέλους. Τώρα, το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Το δικαίωμα πρωτοβουλίας τι σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και την αρμοδιότητα να αποσύρει μία πρόταση και αυτό είναι τμήμα του δικαιώματος ε, πρωτοβουλίας. Η πρωτοβουλία δεν είναι μόνο να καταθέτεις μία πρόταση, είναι και να αποσύρεις μία πρόταση. Έχεις το δικαίωμα. Ε, έχει την εξουσία για τη διαχείριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι την έχουμε ασκήσει αυτή με τον ορθό τρόπο, διότι Αναφέρουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι τμήμα της πρότασης για το 2013 το πρόγραμμα εργασίας. Το συζητήσαμε σήμερα το πρωί και άκουσα με μεγάλη προσοχή όλα τα σχόλια που κάνατε. Αλλά δεν έχει νόημα να μην υπάρχει η δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει μια πρότασή της. Αυτό είναι και κατά των συνθήκων, αλλά και της αρμοδιότητα και τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Εγώ δεν είμαι ούτε εγώ ικανοποιημένο με τη θέση του Συμβουλίου. Προσπαθήσαμε επανειλημμένα να το συζητήσουμε μαζί τους. Ποτέ δεν επέδειξαν την ε, προθυμία ουσιαστικά. Αλλά είναι προφανές ότι δεν πρόκειται το προσεχές διάστημα να βρούμε πλειοψηφία στο Συμβούλιο και αυτό σαφέ είναι. Και ε, δεν ξέρω, ίσως μπορεί η Προεδρία κάπως να μας βοηθήσει. Ποιος ξέρει. Κύριε Λάγκε, κάνετε ερώτηση. Ε, με ποιον είμαστε, με το Συμβούλιο, με το Κοινοβούλιο. Ε, τώρα περί αυτού πρόκειται. Μην τα λέτε αυτά. Εμείς θέλουμε να βρούμε τη σωστή λύση. Και ο κύριος Μορέιρα είπε, μα γιατί δεν αλλάζετε την πρότασή σα κατά τη διάρκεια τη διαδικασία. Μα πραγματικά το εννοείτε τώρα αυτό που λέτε κύριε Μωρέιρα. Εσείς που είστε και εξέχων συνταγματολόγος, κατά τη διάρκεια της ε, ε, διαδικασίας μπορούμε να αλλάξουμε τη νομική βάση, να την ε, ανατρέψουμε τελείως. Μα αν γίνει κάτι τέτοιο, εντάξει, α το μελετήσουμε. Αν, συμβεί, αν υποχρεωθούμε να το κάνουμε, θα πρέπει να καταθέσουμε νέα πρόταση. Βέβαια, απομένει να αποδειχθεί ότι υπάρχει υποστήριξη για αυτή την πρόταση. Αλλά στην τρέχουσα διαδικασία δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν είναι σωστή πρακτική αυτή, θεωρώ. Αν το συζητούσαμε σε πανεπιστημιακό επίπεδο, είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνούσατε στα γαλλικά. Επίσης με, επέκριναν, με για φιλελευθερισμό. Ναι κύριε Ζαντό, φιλελεύθερος είμαι. Εδώ όμως εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο. Δεν εκφέρω την προσωπική μου άποψη, αλλά την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κατά τα άλλα, έχετε καμιά φορά την τάση να συγχαίρετε τον φιλελευθερισμό με τον καπιταλισμό. Δεν ταυτίζονται αυτές οι δύο έννοιες, δεν του παρόντος να τα αναλύσω αυτά. Ε, και έρχομαι σε κάποια σχόλια που έγιναν για τον Μπαγκλαντές και μας λένε μα είναι σκάνδαλο όλο αυτό που συμβαίνει, τα προϊόντα αυτά παράγονται ε, ε, στον Μπαγκλαντές που δουλεύουν αγόρια και κορίτσια για μισθούς πείνας, ελεηνούς και άθλιους και σε συνθήκες τελείως απαράδεκτες. Η αλήθεια είναι αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Και χθε είχαμε τη συζήτηση για τον Μπαγκλαντές. Δυστυχώς ήμουν στο Παρίσι και δεν μπορούσα να συμμετάσχω στη συζήτηση, γιατί ήμουν στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κατά τα άλλα συζήτηση εκεί. This, you know? Αλλά κάτι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ναι, για τον Μπαγκλαντές παράδειγμα. Και πιστεύω ειλικρινά ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερους κανόνες για τις χώρες εκείνες που μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους ε, ελεύθερα και να ε, εισάγουν και ελεύθερα προϊόντα. Το Μπαγκλαντές είναι χώρα στην οποία εξάγουμε τα πάντα πλην όπλων. Ε, δεν ξέρω, ίσως χρειαστούν επιπλέον συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας Ενδεχομένω ένα πρόγραμμα, ο δικό χάρτη, κάτι τέτοιο, σε συνεργασία με την κυβέρνηση όχι μόνο του Μπαγκλαντέ και άλλων κρατών και ευρωπαϊκών εταιριών που έχουν και ευθύνη σε σχέση με όλα αυτά. Είμαι πρόθυμος να το κάνω, αλλά τώρα μην τα αναμειγνύουμε με αυτά σας παρακαλώ. Θα ήθελα να το πω και στον άλλο συνάδελφο. Σας παρακαλώ μην το συγχαίρετε με το παρόν, γιατί τώρα τι γίνεται. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν την ευκαιρία να εξάγουν τα προϊόντα τους στην αγορά μας. Δεν θα έχουν ποτέ τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δική τους βιομηχανία, ούτε την κλωστοεφαντοργία, αν είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται με ακριβώς τις ίδιες συνθήκες με εμά. Αυτές είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και οικονομίες. Εμείς είμαστε μια όρημη οικονομία. Αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά κάποια ελάχιστα πρότυπα και απαντήσεις. Είμαι πρόθυμο να το εξετάσω αυτό, γιατί και εγώ θεωρώ τελείως απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Ε, πρόσφατα αυτή η πυρκαγιά που δεν είναι και η πρώτη, το πρώτο εργοστάσιο που πιάνει φωτιά, το είδα και την περασμένη εβδομάδα. Τι γίνεται στη βυρσοδεψία, εργάζονται με πάρα πολύ επικίνδυνα προϊόντα. Λοιπόν, αυτό τι σχέση έχει τώρα με τη σήμαση προέλευσης. Καμία σχέση. Μην το αναμειγνύετε σας παρακαλώ. αν δεν έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν τα προϊόντα τους στις δικές μας αγορές, τότε ε, είμαστε και προστατευτιστές και δεν είμαστε και ε, ανθρωπιστές. Θα πρέπει να βρεθεί εκεί μια σωστή ισορροπία. Σύντομα, ήθελα να το πω αυτό, Βεβαίως θα επιμείνουμε στην πρόθεσή μας και θα αποσύρουμε την πρόταση. Ε, ενεργά θα εργαστούμε για την υποβολή νέας πρότασης. Είμαι πρόθυμος να το συζητήσω μαζί σας, καθηγητή κύριε Μορέιρα, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, όχι την άλλη εβδομάδα, αλλά σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι το θέμα δεν είναι εύκολο. και για τα εισαγόμενα προϊόντα και για τα χώρια παραγωγής. Δεν ξέρω, ίσως να το επιβάλλαμε μόνο στα δικά μας προϊόντα. Αυτό είναι πιο συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ. Θα γίνουν πολλές συζητήσεις με τη βιομηχανία. Εντάξει. Η δημοκρατία αυτό κάνει, συζητά. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Αυτή δεν είναι καλή. Ε, είναι καταδικασμένη να αποτύχει, ποτέ δεν πρόκειται να περάσει και η μόνη σωστή πολιτική λύση είναι να την αποσύρουμε. Ευχαριστώ. Uh, a conclusion... Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Μετά τη συζήτηση ε, κατατέθηκαν τέσσερις προτάσεις ε, ψηφίσματος. Έκλεισε η συζήτηση και θα